και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 2 ε, το απόγευμα. Και κατόπιν από τις 3 μέχρι τις 11. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές, το διοικητικό προσωπικό και τους διερμηνείς. Και εμείς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Καλό σας βράδυ. Και καλή ξεκούραση ή καλή όρεξη αν κάποιοι που σας πάνε για δείπνο.